Pour le début, nous souhaitons la bienvenue aux membres de la Commission de l'agriculture du Bundestag allemand qui participent aujourd'hui à notre réunion. Et nous passons à l'ordre du jour. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα η έγκριση, δεν υπάρχει καμία παρατήρηση ή ένσταση, επομένως θεωρώ ότι την εγκρίνεται. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε όλες τις γνώσεις ε, ε, εργασίας της συνήθεια της Επιτροπής μας και το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 1ης και 2ης Ιουνίου εναστότος έτου, αλλά και της 8 ης Μαΐου του ιδίου έτους. Έχετε κάτι ε, τώρα ή μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως αλλιώς θεωρώ ότι τα εγκρίνεται. Επίσης σας ενημερώνω ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου, web streaming. Και τώρα, Περνάμε τώρα το άλλο θέμα που είναι Αλυστεί φοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη. 229 τροπολογίες έχουν κατατεθεί και επίσης έχουμε και δύο ε, γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων επιτροπών. Ο δε εισηγητή έχει 17 τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε και έχουν ζητηθεί και καταδίραση ψηφοφορίε. Κύριε Μποβέ, αν θέλετε, δύο λίγων, μπορείτε πριν την ψηφοφορία να μιλήσετε. Μπόβε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω για όλους αυτούς τους μήνες για τη δουλειά τους τους συναδέλφους που μου ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους και πιο συγκεκριμένα για τόσα έγιναν ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και βελτιώσουμε αυτό το κείμενο. Είναι σημαντικό επίσης και το έργο που επιτελέσαμε όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες εκεί που έπρεπε να δουλέψουν από κοινού σκληρά για να ολοκληρώσουμε αυτές τις 17 συμβαστικές τροπολογίες. Όλοι συνέβαλαν, όμως δυστυχώς καταλήξαμε για κάποιες διατάξεις να έχουμε καταδιέρευση φορεία ψηφορία και αυτό είναι κρίμα, διότι είχαν διατυπωθεί συμβαστικές τροπολογίες και προσπαθήσαμε με τη δουλειά που κάναμε να μπορέσουμε πάντα να τα βρούμε όταν ε, ήταν δυνατό επομένως εδώ δουλέψαμε σκληρά ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά το όσα κάναμε για το μέλλον διότι έχουμε την έκθεση Lion όσον αφορά την αναθεώρηση της ΚΑΠ και θέλουμε τώρα να φέρουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και διανομή των σχετικών προϊόντων ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες θετικές πινελιές, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, να υπάρχει καλύτερη γνώση του κόστους παραγωγής και της αλλαγής κάποιων διατάξεων, ούτω ώστε με αυτή την έκθεση να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις για τους ε, αγρότες, για το γεωργικό κόσμο γενικότερα. Με αυτό το πνεύμα κινηθήκαμε. Όσον φροντίζουμε που σήμερα καλούμεθα να ψηφίζουμε, όλους και όλες σας ευχαριστώ για το όσα κάνατε. Νικουλέσκου. Και τώρα πάμε να ψηφίσουμε όσον αφορά τις τροπολογίες. Πρώτη τροπολογία. Τι είναι υπέρ. Qui est contre? Ποιοι είναι κατά. Abstention. Αποχές. Εγκρίνεται. κύριο. Λέει ο πρόεδρος. Πάμε στο 2. Υπέρ. Κατά. Abstention. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Abstention. Rejeté. 7. 6 εγκρίνεται. 7 υπέρ. Abstention. Adopté. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά Αποχές. Για το 8 να κάνουμε επαλήθευση, λέει ο πρόεδρος, και ψηφίζουμε. Πέρασε. Α, η, η κάρτα Δεν πειράζει για μένα να ψηφίζετε κατά, δεν πειράζει που δεν λειτουργήσει η κάρτα, λέει. Για να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Χέσλινγκ, έχετε το λόγο. Τι είναι, έχετε πρόβλημα τεχνικό με την κάρτα. Είπαμε, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία για το 8 ψηφίζουμε. Ah, Πέρασε. Είσαι adopté. Amendement numéro 9. Qui est pour? 9. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Abstention. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Le vote est clos. Et c'est adopté. εγκρίνεται. 11, υπέρ. Κατά. Abstention. Αποχές. Απορρίπτεται το 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά πρέπει να γίνει επαλήθευση για το 14 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 22 κατά αποχές απορρίπτουν. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Εγκρίνεται 24, 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτη της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο, η πρώτη κατά διέρεση χωριστά πρώτα το πρώτο τμήμα. Για την πρώτη τροπολογία της ΣΥΜΚΟ υπέρ. Ποιοι είναι, είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η πρώτη συμβαστική τροπολογία συμπληρωμένη από προφορική τροπολογία του κυρίου Άλβες. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να λάβω το λόγο για να σας πω ότι η λέξη price, τιμή, υπήρχε στο αρχικό κείμενο το οποίο συμφωνήσαμε, αλλά κατόπιν όμως το τελικό κείμενο δεν επαναδιατυπώθηκε, δεν επανασυμπεριλήφθη. Η λέξη τιμή, price. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πενήντα τρία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πενήντα τέσσερα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται

Αποχές. Εγκρίνεται. Η υπερθμόν 16 της ΙΜΚΟ. Υπερ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμβη. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική τροπολογία υπερθμών 3 σε τρία διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 με προφορική τροπολογία. Κύριε Αλβέζη, έχετε το λόγο και πάλι. Θα ήθελα να πω κάτι για να προσθέσω. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κλπ. Πρώτη για αυτή την προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. 89, λέει ο πρόεδρος, δεν, άλλο. 89 κατά αποχές, εγκρίνεται, 89. 91 πει υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 92. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο, 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική υπερθυμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε επαλήθευση το 114 ψηφίζουμε κάποιος ψηφίσει παραπάνω για το ΕΛΚ Θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. ο Πρόεδρος, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα ξανά το 114. Le vote Πέρα Εγκρίνεται και πάμε στην υπαριθμό 6 της ΕΝΒΗ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτε. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτε. Συμβαστική παραθυμών 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική είναι 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμών 7 εις δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν κρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 11 εις δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχέ. Δεν κρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 171. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτονται. Συμβασική τροπολογία υπαριθμών 12. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται Συμβαστική υπερθυμών 13. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 188. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτωση. 190 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μόνο 14 σε δύο τμήματα για το πρώτο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπής περιβάλλοντος, παριθμόν 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περιβάλλοντος, 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200. Υπέρ. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν μεταφράζεται ο πρόεδρος. Στα αγγλικά λένε. Στο 3, στο 3. Βάλτε στη θέση 3 το κουμπάκι για να ακούσετε τη μετάφραση προς τα αγγλικά. Στο τρίτο κανάλι της κονσόλας. Στο τρίτο. Okay. On vote sur l'amendement 200 qui est pour. Ε, είπαμε για την τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές 200 est 201 qui est pour, contre, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 207. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 214 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 215 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Allez, vas-y. 220. 219, c'est quoi C'est refusé quoi 219 est rejeté. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 200... Το 219 απορρίφθηκε, περνάμε στο 220, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 221 υπέρ κατά αποχές δεκτό 222 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 223 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 224 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή και 229 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε με τις κάρτες μας το σύνολο του τροπολογημένου ψηφίσματος. Ξεκινάει η ψηφοφορία.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 Η διευμηνία λειτουργεί πλέον, θα επανέλθω στη γαλλική γλώσσα, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Mm. Το επόμενο θέμα, προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους και λόγους έρευνας, Η συγκήτρια κατάφερε να συμφωνήσει με το Συμβούλιο στο θέμα της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται ε, για επιστημονικούς και ερευνητικού λόγους. Μας έστειλε την άποψή του το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου για να περάσουμε σε μια συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση ο πρόεδρός μας, ο κύριος Δεκάστρο, απέστειλε μια επιστολή στο Συμβούλιο και δεσμεύθηκε να γίνει δεκτή η πρόταση χωρίς τροπολόγηση από την Επιτροπή μας και από την Ολομέλεια. Έχετε το λόγο κυρία Γέγκλε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι διαπραγματεύσεις με την Ισπανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία, για την προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικές έρευνες και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Διαπραγματεύσεις λοιπόν αυτές οδηγήθηκαν σε πέρας και ελπίζω σε αίσιο πέρας να οδηγηθούν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνέχεια, η συνέχεια τους δηλαδή. Και σήμερα με χαρά μου μπορώ να σας δώσω μια επισκόπηση των συμβιβασμών στους οποίους καταλήξαμε στην τελευταία μας συνάντηση τριμερούς διαλόγου στις 7 Απριλίου μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επί της ε, συμβαστικής λύσης που είχαμε βρει ήδη με τη Σουηδική Προεδρία τον Δεκέμβριο του 2009 και να καταλήξουμε σε λύση για τα εκρεμή θέματα μετά από την θέση σε εφαρμογή βέβαια της συνθήκης της ε, Λισαβόνας αυτά τα θέματα ήταν η ε, επιτροπολογία και οι εκτελεστικές διατάξεις και μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε μια λύση για την εφαρμογή τους. Τους μήνες που πέρασαν η νομική υπηρεσία εξέτασε και επεξεργάστηκε νομοτεχνικά την συμβαστική λύση την στην οποία καταλήξαμε. Στις 3 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως σε πρώτη ανάγνωση το συμβαστικό αυτοκείμενο. Θα ήθελα τώρα να πω το εξής το οποίο για μένα είναι σημαντικό. Όλοι οι συνεργάτες των διαφόρων υπηρεσιών, αμφωτέρων των φίλων της νομικής υπηρεσίας, της γραμματείας της Επιτροπής μας, καθώς επίσης οι σκιώδεις και εισηγητές, καθώς και οι συνεργάτες και συνεργάτες των σκιωδών εισηγητών. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά τα πρόσωπα να τα ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουηδικής και Ισπανικής Προεδρίας, καθώς επίσης να ευχαριστήσω όλους τους μεταφραστές που μας συνόδευσαν στη δύσκολη αυτή πορεία, γιατί ήταν και δύσκολο να μεταφραστούν τα κείμενα αυτά. Μετά τώρα από 1,5 χρόνο έχουμε καταλήξει συμφωνία στο δύσκολο αυτό θέμα το οποίο, η οποία λύση που δίνεται θα βελτιώσει την προστασία των ζώων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα θα διατηρήσει την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου όπου διεξάγεται έρευνα. Η ισχύουσα οδηγία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς χρονολογείται από το 1986 με την συμφωνία επιτυγχάνεται ο σημαντικός στόχος να υπάρχουν ενιαίες συνθήκες για την επιστήμη και την οικονομία, ταυτόχρονα να βελτιωθεί η προστασία των ζώων πραγματικά και αυτά βεβαίως να καταστούν απαιτητά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βάση είναι μια τριπλή αρχή της αποφυγής και της, βελτίωσης, της πρόληψης αποφυγής και βελτίωσης εν τέλει των ε, πειραμάτων που χρησιμοποιούν ζώα. Τώρα, θα ήθελα να ε, σας επισημάνω ακόμα μερικά σημαντικά. Στις διαπραγματεύσεις μπορέσαμε να εξετάσουμε και να ταξινομήσουμε όλες τις διαδικασίες ανάλογα με τα δεινά που ε, αναγκάζεται να υποστεί το ζώο και ε, με τη βαρύτητα των ε, δεινών αυτών. Η έγκριση τώρα των πειραμάτων, πειράματα κατά τα οποία χρησιμοποιούνται ζώα δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς πρώτερη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Με άλλα λόγια, ένα σχέδιο έρευνας, ένα project δηλαδή μπορεί να διεξαχθεί μόνο εφόσον μπορέσει να επιτύχει την έγκριση της δημόσιας αρχής και σε ό,τι αφορά την συμβατότητα του project αυτού με την τριπλή αρχή που ανέφερα προηγουμένως. Και πέραν αυτού, επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα και αναδρομικής αξιολόγησης Για το μέγα θέμα τώρα των ε, μεγάλων πυθίκων. Εκεί υφίστανται ε, σαφείς και σημαντικοί περιορισμοί. Σε περιπτώσεις διεθνικής συνεργασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον δεν έχουν γίνει πρώτα οι κατάλληλες έρευνες ε, σε κλινικών συνθήκων για περιπτώσεις όπου, είναι, ε, όπου πρόκειται για έρευνα για φάρμακα τα οποία ενδεχομένως να, ε, από τα οποία ενδεχομένως να κινδυνεύει η ζωή τους. Κάθε χώρα μέλος τώρα οφείλει να ιδρύσει Εθνική Επιτροπή που θα παρακολουθεί την κατάσταση των πειραματοζώων και ό,τι έχει σχέση με την αγορά, διατήρηση, εκτροφή ε, ζώων και που θα εξασφαλίζει η ίδια Επιτροπή και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τα ζώα επιτρέπεται να θανατώνονται μόνο από πρόσωπο με, ειδική εκπαίδευση. Εναλλακτικοί τρόποι θανάτωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εάν δεν ε, οδηγούν σε επιπρόσθετους πόνους. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη υψηλών επίπεδων προστασίας των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για την εκτροφή και διατήρηση των ζώων. Οι δε μεταφορές των ζώων μπορούν να γίνονται πλέον μόνο με τήρηση αυστηρών προδιαγραφών. Εναλλακτικές επιλογές τώρα για πειράματα με ζώα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον αναγνωρίζονται εκ του νόμου. Ο αριθμός των χρησιμοποιημένων πειραματοζών πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν τα μέτρα σχετικά με την εκτροφή και διατήρηση των ζώων, καθώς επίσης και να βελτιώσουν κάθε ε, παράμετρο της χρήσης τους, ώστε οι πόνοι και τα άλλα δεινά τα οποία υφίσταται τα ζώα να περιοριστούν στο ελάχιστο. Επιθεωρήσεις. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό θέμα και εδώ νομίζω πετύχαμε πραγματικά πολλά πράγματα και ιδίω μετά από τη μονή της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κατορθώσαμε να επιτύχουμε την έγκριση ενός αυστηρού συστήματος που προσαρμόζει τον αριθμό ε, των επιθεωρήσεων ε, στον κίνδυνο, στον προβλεπόμενο κίνδυνο. Οι εκτροφείς τώρα μεταφορείς και όσοι χρησιμοποιούν ε, μεγάλους πυθίκους, πρωτεύοντες δηλαδή, ελέγχονται αναέτος. Εφόσον υπάρχουν επιφυλάξεις, η Κομισιόν έχει την δυνατότητα να ελέγχει το σύστημα χορήγησης πληροφοριών των χωρών μελών. και να διεξάγει ελέγχου, να ζητεί να διεξάγονται έλεγχοι μάλλον, απροειδοποιητά. Εν συμπεράσματι, το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφέ οι διαπραγματεύσεις, όπως και στην πρώτη του ανάγνωση τη 5 η Μαου 2009, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ώστε να επιτευθεί ο στόχος της απόλυτης αποφυγής της χρήσης πειραματοζών σε επιστημονικά πειράματα. Αυτός είναι βέβαια μακροπρόθεσμος στόχος. Σήμερα ακόμη δεν είμαστε σε θέση να καταργήσουμε τελείως την χρήση πειραματοζώων. Μετά από 1,5 χρόνο, 1,5 έτος εντατικότητα των συζητήσεων και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν επιτύχαμε και το λέω με πραγματική πεποίθηση, επιτύχαμε να λύσουμε τον δύσκολο αυτό δεσμό, τον δύσκολο κόμπο ανάμεσα σε προστασία των ζώων και σε ε, απαιτήσει των κέντρων που διενεργούν πειράματα. Ώστε να εξασφαλίζεται και η υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και η κάλυψη των αναγκών των πειραματικών κέντρων. Πρόκειται για προδιαγραφέ προστασία των ζώων που έχουν πραγματικά διεθνώ υποδειγματικό χαρακτήρα. Και παρόλα αυτά διατηρεί τον πρωτοπόρο ρόλο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τόπος όπου μπορούν να διεξάγονται πειράματα. Τώρα έχουμε μπροστά μας ε, την συμβαστική λύση του Απριλίου που ενέκρινε στις 3 Ιουνίου το Συμβούλιο χωρίς ψήφους κατά Έρχεται λοιπόν τώρα ενώπιόν μας σε δεύτερη ανάγνωση και καλεί το Κοινοβούλιο ε, να τον εγκρίνει σε ολομέλεια. Οι σκιώδεις ηγητές στην τελευταία συνάντηση του τριμερούς διαλόγου ήδη κατέθεσαν τη σύμφωνη γνώση τους, γνώμη τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας έχει αποστείλει σχετικέ επιστολές στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί της ουσίας τώρα, Τροπολογίε μπορούν να κατατεθούν, το λέω αυτό, διότι οφείλω να το πω, λέω όμως επίσης σαφώς ότι μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει με τους κοιοδησίτες ότι δεν επιθυμούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Η έκθεση θα αποβεί πραγματικά καλή έκθεση εάν μπορούμε όπως έπραξε και το Συμβούλιο, να υποστηρίξουμε ομόφωνα το περιεχόμενο της έκθεσης. Και επιμένω ομόφωνα διότι η ίδια μου η χώρα, η Γερμανία, απέσχε. Όχι τόσο διότι δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά διότι το Υπουργείο, το δικό μας το Υπουργείο Έρευνας, θεώρησε ότι ο συμβασμός δεν είναι επαρκής. Διότι η η Γερμανία περιλαμβάνει στο ε, σύνταγμά της, στο θεμελιώδη της νόμου, την ελευθερία της έρευνας. Το δε δικό μας Υπουργείο Γεωργίας συμφώνησε. Αλλά και η προστασία των ζώων περιλαμβάνεται στον θεμελιώδη νόμο μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δύο πόλοι που και οι δύο περιλαμβάνονται στο ε, σύνταγμά μας προστασία των ζώων και ελευθερία της έρευνας. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό για μας εδώ. Εμείς καταλήξαμε σε καλό συμβασμό. Γνωρίζω για παράδειγμα για την Γαλλία ότι η Γαλλία θα ήθελε <clears throat> πράγματι περισσότερη ελευθερία της έρευνας. Παρ' όλα αυτά συμφώνησε. Γνωρίζω ότι κάτω χώρε θα προτιμούσαν εντονότερη προστασία των ζώων. Παρ' όλα αυτά και αυτές προσυπέγραψαν διότι προτιμούν να διατηρήσουν το καλό αυτό συμβαστικό αποτέλεσμα παρά να αρχίσουν από την αρχή. Γι' αυτό παρακαλώ όλες και όλους να πράξουν πάντο δυνατό ώστε το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας να περάσει από την Επιτροπή μας και μετά στην Ολομέλεια. Θα έχουμε την ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Και εν τέλει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι όλες και όλους για αυτή την εντατικότητα της εργασία των τελευταίων δύο ετών. Ευχαριστώ κυρία Γιέγκλε. Κυρία Εύανς έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιέγκλε Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια Πρόκειται για μια αλλαγή στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία καλούμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα. Υπάρχουν όμως τρία σημεία στα οποία η πολιτική μου ομάδα επιμένει και τα οποία έχει θέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τριμερούς διαλόγου. Θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή σε σχέση με αυτά τα τρία σημεία, τότε η κοινή θέση είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα είναι ασθενές σε κάποιους τομείς και δεν θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε. Στο 2α, σχετικά με τα εθνικά αυστηρά εθνικά μέτρα, η κοινή θέση λέγει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν προς στιγμή τα μέτρα τα οποία ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Εμείς ε, ζητάμε να μπορούν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν επιπλέον ε, τέτοια μέτρα. Να μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια της νομοθετικής διαδικασίας και όχι ένα ανώτατο όριο αν θέλετε. Στο 9.3 θεωρούμε ότι όπου υπάρχει εναλλακτική λύση θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μην απαγορεύεται η χρήση εναλλακτικών λύσεων. Και για το 8, για τα πρωτεύοντα ζώα, η αναφορά στην κατηγορία αυτή των ζώων που δεν, έχουν, που δεν χαρακτηρίζονται από ανθρώπινα κριτήρια δεν έχει γίνει δεκτή στην καινούργια πρόταση και ο Χάσλιπ έχει καταθέσει τροπολογίες για τα τρία αυτά σημεία Έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά πάρα πολύ. Αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η κυρία Γέγκλε, αλλά εμένουμε στις θέσεις αυτές. Κάπουλα Σάντους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο είναι κάτι το οποίο άπτεται και του συναισθηματικού μας κόσμου. Είναι μια προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Είχε ξεκινήσει την προσπάθεια στο προηγούμενο κοινοβούλιο ο τέος πρόεδρός μας ο κύριος Πάρις και το συνεχίζει η κυρία Γέγκλε. Αλλά εμείς μιλάμε περισσότερο από ό,τι φαίνεται για τα δικαιώματα των ζώων παρά για τα δικαιώματα του ανθρώπου αυτό δεν είναι κακό το να ξοδεύουμε δηλαδή πολύ χρόνο στα θέματα των δικαιωμάτων των ζώων. Δεν είναι κάτι το αρνητικό και οι προτάσεις τις οποίες κάνει η κυρία Γέγκλε είναι συνενετικές και θα πρέπει να γίνουν δεκτές. Η πολιτική μου ομάδα θα συμφωνήσει με την πρόταση Γέγκλε και θα την υποστηρίξει και την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει και για το πολύ καλό κλίμα το οποίο κράτησε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Je donne la parole maintenant à Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γέγκλε. Η δουλειά της ε, ήταν εξαιρετική σε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πολύ σπάνια θέματα, που προκαλείται άμεσα το ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια θα συμφωνήσω σε κάποιους τομείς ε, με την ε, κυρία Evans. Η συμβιβαστική πρόταση την οποία έχουμε όμως μπροστά μας, θα ήθελα να πω και στην κυρία Evans, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλήξουμε κάπου. Και εγώ είχα την δυνατότητα να επισκεφθώ την οργάνωση προστασίας των ζώων, το Παγκόσμιο Συμβούλιο μάλλον προστασίας των ζώων, την προηγούμενη εβδομάδα και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τις προτάσεις Γέγκλα και γι' αυτό δεν θα ήθελα παρακαλώ να κατατεθούν τροπολογίες οι οποίες θα έχουν σαν μοναδική επίπτωση την κολυσιεργία και την περαιτέρω καθυστέρηση. Χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία, το πετύχαμε αυτό. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη σύγχρονη επιστήμη και τις ανάγκες της έρευνας από τη μία με την άλλη ε, την αγάπη και την συμπάθεια και την τρυφερότητα την οποία τρέφουμε απέναντι στον κόσμο των ζώων. Ευχαριστώ την κυρία Γέγκλε. Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα των φιλελευθέρων ομόφωνα ή αν όχι ομόφωνα σε μια τεράστια πλειοψηφία θα στηρίξει την πρότασή της. Μπορείτε να κλείσετε κυρία Γέγλε. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες Ήβανς, κυρία Πάουλσεν, κύριε Κάπουλα Σάντος. Γνωρίζω τις ενστάσεις σας Τις έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και της κυρίας Πάουλσεν, η οποία πάντοτε προσπάθησε να προσφέρει υποστήριξη. Βέβαια, περί συμβιβασμού πρόκειται. Δεν υπάρχουν ιδεώδεις λύσεις. Το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Ένα συμβασμό ποτέ δεν μπορεί να έχει ιδεώδη χαρακτήρα. Ούτε άλλωστε φτάσαμε στο τέλος πραγματικά της προσπάθειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βρίσκομαι εδώ από το 1999 ευρωβουλευτής. Σε πόσες περιπτώσεις επετεύθη η πραγματική ανανέωση μιας οδηγίας. Και ειδικότερα τις οδηγίες αυτής, που συχνά πολλοί δεν ήθελαν να την αγγίξουν. Η Κομισιόν εργάστηκε επί του θέματος, το Συμβούλιο εργάστηκε πάνω στην ίδια βάση και αν δείτε μέσα στο χρόνο πόσες ομάδες ανθρώπων ασχολήθηκαν, πόσες ρυθμίσεις έγιναν ε, και ήδη και με το γερμανικό παράδειγμα που σας έδωσα πριν προσπάθησα να καταστήσω σαφές πόσο δύσκολη είναι η θέση του καθενός μας. Αλλά μπορέσαμε πραγματικά από κοινού και βεβαίως και εσείς κυρία Ιβανς, το λέω ρητά, γιατί πρέπει κανείς να προβάλλει τις απαιτήσει, τις αξιώσεις του, ώστε πραγματικά εν τέλει να επιτευχθεί πραγματικός συμβασμός. πραγματικά το μόνο που μένει να πράξω εδώ σήμερα είναι ναι. να ευχαριστήσω και πάλι όλες και όλους και να παρακαλέσω να συνεχιστεί η προσπάθεια να περάσουμε τις δύο αυτές φάσεις που μας μένουν, δηλαδή μια φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το Σεπτέμβριο πλέον στην Ολομέλεια. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας, η οποία γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας μέσα σε αυτό το σύστημα μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αρχίζουμε λοιπόν πραγματικά τώρα με το νέο σύστημα και νομίζω δίνουμε παράδειγμα ε, και στο υπόλοιπο κοινοβούλιο για το πώς μπορεί να εξελιχθεί πιο πέρα αυτή η διαδικασία. Πριν κλείσει η συζήτηση, πάρα πολύ σύντομα ένας τελευταίος ομιλητής. Θα είμαι πράγματι πάρα πολύ σύντομο. Το θέμα αυτό, λέει ο κύριος Νίκολσον, έχει ξεκινήσει να συζητιέται ήδη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και ο κύριος Πάρη ήταν υπεύθυνο. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γέγκλε για την τεράστια προσπάθεια που έκανε σε έναν τομέα ο οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να φτάσει θα έλεγα στην μέγιστη, θα έλεγα, στο μέγιστο βαθμό συνένεσης που μπορούμε να πετύχουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τις προτάσεις αυτές, δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Ας πάρουμε πια αυτή την απόφαση τώρα, γιατί όπως είπα η συγγήτρια έκανε μια τεράστια προσπάθεια για να πετύχει τους συμβιβασμούς. Προφανώς συμβιβασμός δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, αλλά όσοι, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε το πετύχαμε. Θα διακόψουμε τώρα την συζήτηση μέχρι τις 4 και 4 όπου θα έχουμε μία συνάντηση με την ε, Ισπανίδα Υπουργό Περιβάλλοντος και Υπέθρου, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου.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 Bonjour de nouveau. Je souhaite la bienvenue à Madame Elena Espinosa, présidente. Συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα την ε, Υπουργό Περιβάλλοντος και μέσω της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Θα μας εξηγήσει πώς έχουν το πράγμα. Nessuna spiegazione, benvenuti. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Σπινόζα. Η πόλη μου από τον νότο της Ιταλίας παράγει εξαιρετικά κεράσια. Δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω προφορικά, σας τα προσφέρω να τα δοκιμάσετε μαζί με την ομάδα προώθησης των οποροκυπευτικών της πόλης μου. Είναι τιμή μας που σας τα προσφέρουμε. Εμείς προσπαθούμε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυηθούμε την ανιχνευσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων τα οποία καταλήγουν στον καταναλωτή σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Είμαι πολύ υπερήφανος που σας παρουσιάζω αυτά τα ωραία φρούτα σε εσά και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και Σιλβέστρης. Merci beaucoup. Η Υπουργό θα μας παρουσιάσει τώρα τον καρπό των προσπαθειών της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της Γεωργίας. Για την ΚΑΠ μετά το 2013, ορίζον 2020, ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας και ανταγωνιστικότητα γενικά του αγροτροφημικού τομέα. Το Μάιο είχαμε, είχαμε οργανώσει μια ακρόαση συγγνώμη, γύρω από τα θέματα αυτά. Είναι θέματα τα οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή μας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα κύριε και κυρίες βουλευτές. Πριν αρχίσω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλβέστρης για αυτό αυτό το, το, ότι φρόντισε να μπορούμε να δούμε από κοντά πόσο ποιοτικά γεωργικά προϊόντα έχουμε. Ήρθα εδώ στην Επιτροπή για να σε όσον αφορά έναν απολογισμό των πεπραγμένων της Ισπανικής Προεδρίας και όσα διαμήφθηκαν στο Συμβούλιο Γεωργίας. Όπως γνωρίζετε, πρώτη για την τέταρτη φορά που ανέλαβε η χώρα μου την Προεδρία. Όμως, κατά το εξάμεινο αυτό, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο εξάμεινο προηγουμένης προεδρίας, είχαμε την θέσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέλαβε καθημερινά καθημερινό της κανονικά παρά μόλις τέλη Φεβρουαρίου. Οπότε και από πλευράς Γεωργίας το έργο μας γίνεται επί τη βάση της διαδικασίας της συναπόφασης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του εξαμήνου της Προεδρίας μας, αλλά και εγώ θα πρέπει να σταθώ σε αυτό το τελευταίο σημείο, μια που Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την καινούργια μέθοδο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να έχουμε μια καινούργια αρχή, μια καινούργια διαδρομή, μια καινούργια όθηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση στα ευρωπαϊκά πράγματα, διότι οι μέλουσες αποφάσεις οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν θα αποκτήσουν περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα. Και όλα αυτά θα, θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις ε, προσδοκίες των Ευρωπαίων. Για να δούμε τώρα τι έχουμε όσον αφορά περισσότερο την ουσία. Θα πρέπει να σας αναφέρω ε, μια, μια, μια σύγκριση. Κάτι το οποίο αφορά αυτό το οποίο συζητήσαμε όταν ήρθα να σας δω τον Φεβρουάριο. Είχαμε πει ότι το έργο μας όσον αφορά πολιτική θα εστρέφει γύρω από τα διατροφής και την υγειοργία θεωρώντας ότι πρόκειται για ε, θέμα στρατηγικής μας για την Ευρώπη. Και γνώρισα από κοντά το έργο του Κοινοβουλίου και τη της Επιτροπής αυτό το εξάμεινο τώρα μπόρεσα να καταλάβω καλά ότι το μήνυμα το οποίο στείλαμε ε, ήταν ένα μήνυμα το οποίο το έλαβε όλη η κοινωνία. Το Δε Συμβούλιο Γεωργίας, το οποίο είχα την τιμή να προεδρεύσω κατά το εξάμεινο, αλλά και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο όλοι γνωρίζουμε ότι το διακύβευμα εδώ είναι το μέλλον της Γεωργίας. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ακριβώς τι κάναμε από πλευρά της Ισπανικής Προεδρίας. Πρώτο πρώτο, το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται όπως και άλλοι τομείς οικονομική δραστηριότητας από αυτή την χρηματοπιστωτική κρίση η οποία έχει χτυπήσει πάρα πολύ σκληρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υπάρξει μια ε, συνολική αντιμετώπιση μέσω της στρατηγικής ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν του 2020 ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα για να μπορούμε να έχουμε επίση ε, ένα, ένα μέλλον βιώσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε διέξοδο στο αδιέξοδο αυτή τη κρίση. Βέβαια δεν ήταν δυνατόν να μην καλύψει τα 2020 και την ε, γεωργική πολιτική. Έτσι θεωρούμε ότι έχουν τα πράγματα και έτσι Νομίζω ότι το βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, οπότε έχουμε αυτές μας τις δεσμεύσεις, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα των ε, Συμβουλίων του, του, του και του Ιουνίου. Οπότε εκεί ρητός αναφερόμαστε στην συμβολή της Γεωργίας και συγκεκριμένα της κοινής αγροτικής πολιτικής ή στους στόχους και τις προτεραιότητες ε, της στατικής για το 2020. αναλάβαμε τη σχετική πρωτοβουλία. Θελήσαμε να αναλύσουμε τη συμβολή της Γεωργίας και της ΚΑΠ στην στρατηγική 2020 οπότε και υπήρξαν δύο συζητήσεις στα Συμβούλια Γεωργίας. Η πρώτη συζήτηση έγινε τον Μάρτιο. Η, η άλλη συζήτηση έγινε στο άτυπο Συμβούλιο της Μέριδα. Βεβαίως προηγήθηκαν πάρα πολλές συναντήσεις με κρατημέλη και με του κλάδου. Οπότε, σε αυτή την προσπάθειά μας βοήθησαν όλα τα κρατημέλη, αλλά και οι εκπρόσωποι των ε, γεωργικών φορέων. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, οργανώσεις νέων γεωργών, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας. Και αυτό το εξάμεινο επίση μπορούσαμε να σημειώσουμε βήματα προόδου όσον αφορά την αναθεώρηση τη ε, διαχείριση ε, τη ε, αγορά και επίση όσον αφορά την αντιμετώπιση τη κρίση αλλά και το ευμετάβολο των τιμών. Οπότε μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια σε κάποια συμπεράσματα και μπορούσαμε επίσης έτσι να εμπλέξουμε και την υπόλοιπη Τρόικα. Δηλαδή το Βέλγιο και την ε, Ουγγαρία. Έγινε επομένω μια προσπάθεια κατά αυτό το εξάμεινο, ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε στο μέλλον να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία να είναι δυνατόν να έχει μια, μια, μια, μια χάραξη πιο μακρόπνοια το 2013. Διότι αναγνωρίζετε και ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να είναι ισχυρή αυτή η πολιτική και να είναι επαρκώ προοικοδοτημένη. Για μας ε, ήταν μεγάλη ικανοποίηση το ότι μας βοήθησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως ε, αυτό εδώ το κοινοβούλιο, αλλά επίσης και ο Παύλο Δεκάστρο, πρόεδρος, όσον αφορά την αναγνώριση του στρατηγική, της στρατηγικής σημασίας της γεωργίας, μια που συμβάλλει πάρα πολύ στην ε, οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση, όπως επίσης και ίστο να διατηρείται η οικονομική δραστηριότητα στην Ήπεθρο να μένει και ο κόσμος. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση της διατροφής με έναν τρόπο αηφόρο, με έναν τρόπο αξιοπρεπή όσον αφορά και τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Οπότε, και εμείς με μεγάλη μας χαρά συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία από πλευρά της δικής σας επιτροπής. Ε, και πάνω στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ ήταν ε, η έκθεση Lion, η Lyon, ε, η οποία έκθεση συμφωνεί με τους στόχους του Συμβουλίου και εμείς θα συνεχίζουμε επομένω το έργο μας με αυτή την αφετηρία, στη συνεργασία μαζί σας και ελπίζουμε ότι αυτό το κείμενο πρόκειται την επόμενη εβδομάδα να εγκριθεί. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι αυτά είναι εύκολα. Όμως, θυμηθείτε πριν από έξι μήνες, τι λέγαμε εδώ. Λέγαμε ότι είναι μια αναγκαιότητα η κοινή γραφική πολιτική να καλυφθεί από την στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιση του 2020. Σήμερα δε ευτυχώς ο στόχος αυτός επετεύχθη και επιμένω ότι πρόκειτο για δύσκολο έργο, αλλά ενεπλάξαν και βοήθησαν πάρα πολύ και προς κάθε πλευρά δεν μπορώ παρά να πω ευχαριστώ. Δεύτερη προτεραιότητα την οποία τάξαμε ήταν το πώς θα βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας αλλά και της ε, διατροφικής βιομηχανίας. Σε πάρα πολλά θέματα ε, δουλέψαμε αυτό το εξάμεινο και η βελτίωση της λειτουργίας της διατροφικής αλυσίδας ε, έγινε κυρίως όσον αφορά την διαφάνεια, όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, όσον αφορά την ενίσχυση των ε, οργανώσεων, των παραγωγών και των ε, άλλων συναφών κλάδων. Σαν αποτέλεσμα των συζητήσεων καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα της Προεδρίας όπου τονίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, σχέσεις ε, σταθερές. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλη αυτή τη διατροφική αλυσίδα και να τονιστεί ότι θα πρέπει ο αγροδιατροφικός τομέας να αναβαθμιστεί. Και για άλλη μια φορά συμφωνούμε. Κατά αυτό το εξάμεινο κάναμε αυτά τα τρία σεμινάρια όσον αφορά τα θέματα της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και νομίζω τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Επίση, θα πρέπει να σα εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση τη εκθέσεω βεβαίω όσον αφορά τη βελτίωση τη ε, λειτουργία, τη ε, παραγωγή, και διανομή των ειδών διατροφή στην Ευρώπη που εγκλήθηκε. Ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο συζητήθηκε ευρέω καθ' αυτό το εξάμεινο ήταν η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής. Τα εξαχθέντα συμπεράσματα κατόπιν αυτών των σχετικών εργασιών και συζητήσεων συζητήθηκαν σαν σημείο α στο Συμβουλίο Υπουργών ε, αύριο. Θα εγκριθούν αύριο, Και αυτό μια που έχουμε συσπηρώσει τα κρατημέλη γύρω από μια συνένεση για το θέμα αυτό και επίσης και αυτόν τον τρόπο θα έχουμε εγγυήσεις ποιότητα στην παραγωγή. Και αυτό θα γίνει με κάποια μέσα και εργαλεία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι το πρότυπο αυτό το ευρωπαϊκό θα έχει αυτή την προσθέμενη αξία που να μας προσδίδει ανταγωνιστικότητα. Επίσης θα πρέπει να αγνοούμε το ότι οι ευρωπαϊκοί τεχνικοί κανόνες θα πρέπει να έχουν και κάποιο είδους προηγούμενη επιστημονική αξιολόγηση και επίσης και με κάποια μελέτη να συνοδεύονται μελέτη οικονομικών επιπτώσεων. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς τα συστήματα επικοινωνίας θα είναι δυνατόν να φτάνουν αυτά τα στήματα επικοινωνίας μέχρι τους καταναλωτές τους ώστε να είναι δυνατόν η προσπάθειά μας η παραπάνω να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Και όπως ο προηγουμένος η ισότητα των φίλων για μας είναι μια προτεραιότητα για όλες τις πολιτικές και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας επίσης προσπαθήσαμε να είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαριστεί. Επίσης θέλουμε η Ήπεθρος να ενισχυθεί επίσης να βοηθούν οι γυναίκες εκεί, να μείνουν εκεί γιατί έτσι η προεδρική δραστηριότητα είναι εξασφαλισμένη. Κατά την Προεδρία μας επίσης θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε τις εργασίες μας και στα θέματα ισότητας των δύο φύλων, κάτι το οποίο για πρώτη φορά συζητήθηκε σε Συμβούλιο Γεωργίας στην Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θεωρεί σωστό η, ισότητα να αποτελέσει αντικείμενο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Φυσικά θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι έχετε αναλάβει να στέξετε κάποια έκθεση γι' αυτό. Επίσης ευχαριστούμε διότι μας δόθηκε η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις βασικές καθητήρες γραμμές του έργου μας και νομίζω ότι η ανταλλαγή των απόψεων πάντοτε ε, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να παρέψουμε επίση να σα πούμε τι άλλο καταφέραμε αυτό το εξάμεινο. Όπω το ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε καινούργια όθηση στην πολιτική απλούστευση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδίω όσον αφορά την conditionalité. Conjunto para aprobar las medidas en favor de las regiones. Για την ερεσιμότητα δηλαδή, επίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε τις ε, περιφέρειες και περιοχές της απότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα γίνει και θα εγκριθεί σαν μέτρο αύριο στο Συμβούλιο, μια που ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ βασικό θέμα της πολιτικής γεωργίας και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε είναι θετικά, και είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο με τον επιτέλεσαμε το έργο μας από τις θέσεις αυτής της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία τόσο σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπουργό, αλλά και ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου ελπίζω να κάλυψα τις ε, προσδοκίες της δικές σας και των Ευρωπαίων. Εν θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής σας που έχουν λάβει μέρος σε όλες αυτές τις συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Εδώ, κάπου αλλού στην Ευρώπη ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Επίρου. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Και οπότε θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε όσον αφορά τις κοινέ μας επιδιώξεις στα πλαίσια της επόμενης Προεδρίας, της Βελγικής, στα πλαίσια της ε, συνεργασίας της Τρόικα των Προεδριών. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο συμφωνήσαμε με Ουγγαρία και Βέλγιο. Και αυτό θα το δείτε τις αμέσως επόμενες μέρες γιατί θέλουμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί με όλους σας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή Έλενα. Σας ευχαριστώ για ένα εξαιρετικό εξάμεινο κατά τη διάρκεια του οποίου προεδρεύσατε. Έγιναν πολύ σημαντικά βήματα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ότι χαρακτηρίστηκε όχι μόνο από το Συμβούλιο Γεωργίας αλλά και περιβάλλοντος και αλληλείας τρία πολύ σημαντικά συμβούλια που δείχνουν τη δουλειά την οποία έχει πετύχει. Ευχαριστώ επίσης για τις στενές σχέσεις που είχες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα έπαιζε στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση στο ανεπίσημο α συμβούλιο στη Μερίδα και νομίζω ότι το εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον χορό των ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Θεώρησα ότι ω συνήθω πρώτα μιλήσουν οι συντονιστέ. Τόσο δεν πειράζει. Και πάλι ευχαριστούμε. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσουμε την απερχόμενη Προεδρία, την κυρία Υπουργό που ήρθε σήμερα, όπως έχει έρθει και άλλες φορές κατά αυτό το εξάμεινο, για την αλήθεια ότι κατέβαλε προσπάθεια να έρχεται σε όλες τις ε, συναντήσεις που κάνουμε και όχι μόνο στην αρχή και στο τέλος. όντως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ισότητα ανδρών γυναικών ε, όσον αφορά το τι γίνεται στην Ήπεθρο γιατί και οι άντρε και οι γυναίκε επιτελούν σημαντικό έργο. Δυστυχώ. υπάρχουν ε, περιορισμοί όσον αφορά την πρικοδότηση κάποιων μέτρων γιατί έχουμε την γνωστή οικονομική κρίση. Πάντως νομίζω ότι αυτά τα οποία λέμε τώρα θα αποτελέσουν ε, ένα, ένα κρατούμενο, θα αποτελέσουν κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσουν να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Επομένως ήταν σημαντική παρουσία της και Υπουργού, αλλά πρέπει να δούμε πού δεν συμφωνούμε. Πρώτα απ' όλα τι όσον αφορά το μέλλον της ε, ΚΑΠ μετά το 2013. Τι θα γίνει με την κοινή πολιτική στο μέλλον, τι θα γίνει με τις άμεσες ενισχύσεις, τι θα γίνει με τον δεύτερο πυλώνα. Γιατί τι θα γίνει, θα έχουμε έναν ή δύο πυλώνες. Ε, μας προβληματίζει η θέση του κόμματός σας. Αυτά τα έχετε πει σε διάφορα χρήματα, σε διάφορα, διάφορα έγγραφα του Υπουργείου σας, αλλά ε, μας, απασχολεί. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει εν ώψη του πώς θα δημορφωθεί κάποιος στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση απόψεων μεγαλύτερη στο Συμβουλίο. Δεν το παλέψατε αρκετά γιατί Σουηδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία είναι χώρες ας πούμε, ας πούμε παίρνουμε που έχουν μεγάλες διαφορές στις προσεγγίσει στα συμφέροντά του. Επίσης ούτε συμφωνούμε μαζί σας ε, ε, όταν λέτε ότι η στρατηγία του 2020 είχε σημαντικές επιπτώσεις. Ότι όλες οι κοινέ πολιτικές ΚΑΠ και συνοχής είναι πολιτικές που θα πρέπει να καλυφθούν από την αρχή του 2020. Δεν συμφωνούμε. Επίσης, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνετε περισσότερα πράγματα για τη γεωργία. Τίποτα δεν καινούργιο δεν πρόκυψε. Τι έγινε με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες δεν έκανατε τίποτα καλύτερο για τις ε, εισαγωγές από τέτοιες χώρες όπως με το Μαρόκο. Υπήρξε αυτή η συμφωνία με το Μαρόκο που δεν μπορούσατε να την κλείσετε. Οι Γεωργοί τι θα κάνουν σε τις χώρες όταν έχουν αρχίσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Τι γίνεται με την ασφάλιση του εισοδήματος. Είναι πάγιο αίτημα αυτό των Ισπανών γεωργών. Τι θα γίνει, υπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις του, ε, του, του Υπουργού. Καπούλα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό. Θα ήθελα όχι μόνο να την ευχαριστήσω αλλά και για να τη συγχαρώ για την εξαιρετική τους δουλειά. Παρακολουθήσαμε προσεκτικά τα επιτεύγματα της Προεδρίας και μπορώ να πω ότι η στάση μας απέναντι στα πεπραγμένα της Ισπανικής Προεδρίας είναι ιδιαίτερα θετική. Όχι μόνο γιατί αρκετά πράγματα τακτοποιήθηκαν, αλλά γιατί η Ισπανική Προεδρία ήταν διαθέσιμη πάντα και έδειξε πνεύμα συνεργασίας, συναντήθηκε μαζί μας επανειλημμένα. Χρειάστηκε να κάνετε ακόμα και προσωπικές θυσίες για να μπορέσετε να κρατήσετε στενή αυτή την επαφή και αντίστοιχη επαφή κρατήσατε επίσης και με τις οργανώσεις των Ευρωπαίων Γεωργών οι οποίοι θεωρούν και αυτή την Προεδρία σας εξαιρετική. Ο ρόλος λοιπόν της Ισπανικής, που έπαιξε η Ισπανική Προεδρία ήταν καθοριστικός ε, σχετικά με το θέμα της γεωργίας και τη στρατηγική του 2020. Δεν μιλάμε πάρα πολύ για τη γεωργία όταν μιλάμε για το 2020. Μιλάμε λίγο, ανεπαρκώς. Αλλά θυμίζω ότι πριν λίγους μήνες δεν μιλούσαμε καθόλου για την γεωργία στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Ήδη λοιπόν αυτό που πετύχατε είναι σημαντικό. Ξεκινήσατε μια πραγματική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και αυτό κάτω από όρους θα έλεγα οι οποίοι ήταν απρόσμενα θετικοί. Τέθηκε η συζήτηση με υπερεθνικό τρόπο προσπαθώντας να γίνουν σεβαστά κυρίαρχα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με μονομένα συμφέροντα κρατών μελών τη διεθνή σκηνή. Σας ευχόμεθα καλή τύχη από εδώ και πέρα στην πολιτική σας προσπάθεια και ελπίζω επίσης και η Ισπανική ομάδα στην Νότια Αφρική ε, να μην είναι τόσο καλή όσο εσείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ Λουίς. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα, ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και για την εργασία που επιτελέσατε στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή συχνά εργαζόμαστε διακομματικά με γνώμονα την ουσία και θέλουμε πραγματικές αποφάσεις επί της ουσίας. Βέβαια ομολογώ ότι δεν βλέπω πολλές θετικές αποφάσεις ουσίας για τη γεωργία στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Μιλήσατε για την στρατηγική του 2020 θα με ενδιέφερε να ακούσω από εσά ποια είναι τα θετικά στοιχεία τα οποία επιφέρατε εσείς στην στρατηγική 2020 ως Ισπανία που είσαστε μια μεγάλη χώρα μέλος και για την στρατηγική του 2020 η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα με σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα πολύ να δω η χώρα σας να παίξει ένα σημαντικό θετικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής. Από τις δηλώσεις σας δεν άκουσα τίποτα εάν θα υπάρξει δηλαδή ισχυρός πρώτος πυλώνας, δεύτερος πυλώνας, συγχρηματοδότηση. Ίσως μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια στο τέλος όταν θα ξαναλάβετε τον λόγο. Μιλήσατε για την ε, προώθηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των τροφίμων. Συμφωνώ μαζί σας. Άλλωστε σήμερα ψηφίσαμε θέλουμε με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε την θέση της οικονομίας. Και αυτό είναι σημαντικό να διασφαλιστεί. Αυτό που θα παραμείνει στην μνήμη μας ως αρνητικό είναι ότι ξανά άνοιξαν οι διαπραγματεύσεις Μερκοσούρ και αυτό μας ανησυχεί πολύ διότι η αγροτική πολιτική μετά το 2013 την οποία συζητούμε και θα συζητήσουμε ακόμα στη διαδικασία συναπόφαση με το Συμβούλιο τους επόμενους μήνες, θα επιτύχει μόνο αν υπάρχει και κάποια προστασία προς τα έξω. Τώρα με τις συμβάσεις Mercosur, εάν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις προδιαγραφές μας ποιότητας, προδιαγραφές προστασίας καταναλωτού, προδιαγραφές προστασίας των ζώων, τότε η προσπάθειά μας αυτή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας δεν θα επιτύχει. Θα παρακαλέσω λοιπόν ειδικά εσάς και την Ισπανία στις διαπραγματεύσει αυτές με τις χώρες Μερκοσούρ καθώς και σε όλες τις διμερείς διαπραγματεύσει, να υπερασπιστείτε το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο. Εάν μπορείτε να μας το υποσχεθείτε αυτό για το μέλλον θα με ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά τα σχόλια σας ευχαριστώ για την συνεργασία Όλοι βέβαια χρειάζεται να συμβάλλουμε για να εξευρεθούν εύλογες λύσεις υπέρ των Ευρωπαίων Γεωργών. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Γκαρσία Περές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρχίζω ευχαριστώντας, κύριε Υπουργό, που σήμερα ήρθε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε επίση για τα όσα έκανε κατά την Προεδρία. Όσον αφορά την ε, παγωτική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξη τη υπαίθρου. Μια που ήταν πολύ κρίσιμη αυτή η καμπή και όσα συζητήσαμε για το Συμβούλιο, για το όσα συζητήσαμε εμεί εδώ, για το μέλλον της ΚΑΠ, νομίζω ότι όλα αυτά βοήθησαν στο να υπάρχει περισσότερη βεβαιότητα στον κλάδο, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να μην υπάρχει αβεβαιότητα. Γιατί, όπως υδρώ το κλίμα, δημιουργείται αγώνια για το μέλλον τους. Άρα το έργο το οποίο επιτέλεσε η Προεδρία και προσπαθώντας μαζί μας να έχουμε βάσεις, διάλογο για την χάραξη της πολιτικής της Γεωργίας το 2013 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τώρα η ώρα για αντιπαραθέσεις, ούτε για να δημιουργούμε μεγαλύτερες αβεβαιότητες από αυτές που ήδη σοβούν στον κλάδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο να στείλουμε, όπως και το Συμβούλιο στον κόσμο, ένα αντίστοιχο μήνυμα ότι η κτηνοτροφία και η γεωργία θα υπάρχουν και στο μέλλον. Και να μπορέσουμε όλα αυτά να εντάξουμε και στην πολιτική για το 2020. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα πάρα πολύ καλά τα πήγε η Προεδρία στο Συμβούλιο, πάρα πολύ καλή ήταν και η συνεργασία μας μέσω του Προέδρου μας και των άλλων συναδέλφων οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και που μιλήσαμε για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε χωρίς να συζητήσουμε για το πώς θα βοηθήσει κτηνοτροφία και γεωργία. Άρα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και είναι κάτι βασικό. Η γυναίκα και η πέτρος. Επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είχα την τύχη να βρεθώ σε μια τέτοια ε, συνάντηση και όλοι συμφώνησαν για τον ρόλο της γυναίκας όσον αφορά το μέλλον της υπαίθρου. Άρα θα πρέπει και εμείς να απασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό και να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι πρέπει, να ληφθούν κάποια μέτρα, εγγύησεις για τη γυναίκα στην Ήπεθρο ευκαιρίες, ισότητα των ευκαιριών. Και επίση κατά κατακλείδα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Τρόικας, δηλαδή το τι θα κάνει στο μέλλον το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Θα πρέπει να είναι προσπάθειες κοινέ. Άρα όχι μόνο δεν χρειάζεται αντιπαράθεση, αλλά χρειάζεται να δείξει κανείς στους ε, Ευρωπαίους γεωργούς, σε όλο τον κλάδο, στο ότι είναι δυνατόν αυτό το οποίο κάνουμε εδώ να γίνονται και στο επόμενο εξάμεινο ε, πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, λίγο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για σημαντικά πράγματα στη διάρκεια της ε, παρεμβάσεώς σας. Μιλήσατε για τον τομέα των τροφίμων, είπατε ότι είναι κρίσιμος για το μέλλον της Ευρώπης, μιλήσατε για ε, βιώσιμη ανάπτυξη, μιλήσατε επίσης για ολοκλήρωση του τομέα. Μιλήσατε για το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής και ότι έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Αυτά όλα και εμένα με απασχολούν πολύ. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε μου να θέσω μια ερώτηση. Έχουμε περιορισμούς. που επιβάλλονται από την Αργεντινή στις εμπορικές συνδιαλλαγές της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι η θέση ή ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ας πούμε να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ. Τρεις ημέρες μετά από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, η Αργεντινή επιβάλλει αυτές τις περιοριστικές αποφάσεις με ευρύ χαρακτήρα. Γνωρίζουμε ότι αρχές Ιουλίου θα είναι ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων. Θα θέλαμε να τηρούμαστε ενήμεροι των προόδων αυτών των διαπραγματεύσεων. Ακούμε τώρα ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα περιστραφούν γύρω από τεχνικά θέματα. Ακούσαμε έτσι στην αρχή. Ακούμε τώρα όμως ότι δεν θα είναι απλώς τεχνικού χαρακτήρα. Έχω την εντύπωση ότι παρετούμεθα από τα δικαιώματά μας. Αντιλαμβάνομαι ότι το εμπόριο πρέπει να απελευθερωθεί, αλλά όχι όμως να οδηγήσει σε ζημία της γεωρικής μας παραγωγής. Εν πάση περιπτώσει, οφείλετε να προστατεύσετε τους γεωργούς ή τουλάχιστον να συνομιλήσετε μαζί τους, να τους εξηγήσετε για ποιο λόγο λαμβάνονται τα μέτρα που λαμβάνονται. Έχω την εντύπωση ότι αυτά γίνονται εν κρυπτό και παραβίστο και ότι ορισμένα μέτρα εισάγονται, θα έλεγα, από την πίσω πόρτα. Αυτά δεν μου φαίνονται σωστά, διότι έτσι εκ προθέσεως βλάπτουμε τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα. Και επίσης είπατε εσείς η ίδια ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής διασφαλίζει τον ανταγωνιστικό της χαρακτήρα. Χρειαζόμαστε κάποια σταθερότητα όμως στην πολιτική αυτή. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι αντιδρούμε σπασμωδικά. Λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα σε απήχηση των όσων διαπραγματευόμαστε με τη Μερκοσούρ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τα όσα κάνατε και για το τι ήρθατε να μας δείτε με μεγάλη μου χαρά πάντως. Είδαμε ότι κάνατε πολλά και φυσικά και, και εγώ άριστο κρίνω το έργο σου όπως και ο κύριος Καμπούλας Σάντος θα, ήθελα να σας πω και εγώ τα ίδια αλλά δεν μπορώ να πω και σαν τον Καμπούλας Σάντος αλλά δεν ξεγελιέται ο κόσμος και η Γεωργή γιατί ε, δεν είναι η Γεωργία για την κυβέρνηση της Ισπανίας. Η Γεωργία ούτε ήταν για την, ε, ούτε, πώς ήταν για την κυβέρνηση της Ισπανικής, δεν ήταν για την προεδρία σας. Χάσατε μια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσουμε όσον αφορά τα αυτά που χρειάζεται ο στρατηγικός αυτός κλάδος. Χρειάζεται δεσμεύσεις, χρειάζεται συστράτευση για το μέλλον. Είπατε για την απότερη περιφέρεια της Ένωσης, είπατε ότι είναι σημαντική η έκθεση αυτή και μιλήσαμε για το μέλλον αλλά πολλές φορές αυτό δεν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Μας είπατε τι κάνατε, αλλά δεν μας είπατε τι δεν κάνατε. Θα ήταν ακόμα πιο ε, υπερήφανη Προεδρία αν είχε κάνει κάτι όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες ελευθέρας, ελευθερό εμπορίο. Ε, ήρθε εδώ ο Υπουργό Εσωτερικών, αλλά πού πήγε ε, το Υπουργείο Γεωργία, τι έγινε με την Κολομβία και το Περού, τα όσα γίνανε εκεί. Από τα 176 πήγαμε στα 70 ευρώ όσον αφορά την τιμή της μπανάνας εκεί. Δηλαδή οι εξελίξεις στην αγορά της μπανάνας ήταν καταστροφικές για την Ευρώπη. Οπότε κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι έγινε, πού ήταν το Υπουργείο Γεωργίας, τι έγινε με το Μερκοσούρ, όλα ήταν αρνητικά. Όχι μόνο για την κτηνοτροφία, γενικά για τη Γεωργία. Πού ήταν το Υπουργείο Γεωργία όταν είχαμε αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε με το Μαρόκο. Μιλάμε για κάποιε συμφωνίε οι οποίε κατέληξαν οι διαπραγματεύσει του σε πάρα πολύ αρνητικέ συνέπειε για του Ισπανού Γεωργού. Επίση, η διαμόρφωση τη τιμολογική πολιτική επίση ήταν πάρα πολύ κακή ε, και, και ξέρουμε ότι έχει επιληθεί και Όλαφ ε, σε κάποιες στον τρόπο διαχείρισης αυτών των συμφωνιών. Γι' αυτό σας λέω ότι υπήρξε μια ευκαιρία που τη χάσαμε. Γιατί ούτε στη Γεωργία ε, μπόρεσε να λάμψει η Ισπανική Προεδρία. Επομένως, ε, όσα δεν κάνατε σαν κυβέρνηση, δεν μπορούσατε να τα κάνετε και σαν Προεδρία. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι ήδη συνεχάρισαν την κυρία Υπουργό. Ήταν έξι μήνες ιδιαίτερα παραγωγική για τον κλάδο που μας ενδιαφέρει. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η προσπάθεια την οποία ανέλαβε η Ισπανική Προεδρία. Μέσα σε έξι μήνες κατάφερε να διατυπώσει αλλά και να θέσει σε εφαρμογή ορισμένες τουλάχιστον από τις ιδέες της πείθοντας τα υπόλοιπα 26 κράτη. Είμαι νέος βουλευτής εγώ εδώ και η Λετωνία την οποία εκπροσωπώ είναι και αυτή μία από τις πιο πρόσφατες χώρες μέλη. Υπογραμμίζω όμως ότι όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναφερόμαστε συχνά στις ενέργειες της, ε, της κυβέρνησης της χώρας μας. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αυτά τα οποία θα περίμενε κανείς να κάνουν ακόμα και όταν υποχρεούνται από το κοινοτικό πλαίσιο. Και πολύ συχνά το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται είναι ότι οι κυβερνήσεις επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους και έτσι δεν καταφέρνουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη κοινοτική πολιτική. Ο παραγωγικός τομέας που μας ενδιαφέρει στην χώρα μου είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Μου είπανε συζητάτε για το 2013, για τη Γεωργία 2020, το 2020, αλλά δεν κάνετε τίποτα για, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι Γεωργοί σήμερα. Ακούμε από τη μία ότι 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και ταυτόχρονα εσείς επιβάλλετε μια ολόκληρη σειρά, ε, θα έλεγα, καταπιεστικών σε εισαγωγικά μέτρων που οδηγούν στη μείωση της γεωργικής παραγωγής. Γιατί σαν παράδειγμα οι άμεσες πληρωμές να συνδέονται με την τελική παραγωγή. Η κατάσταση στη χώρα μου είναι ιδιαίτερη είναι αλήθεια. Γιατί έχουμε εδάφη προς καλλιέργεια τα οποία ακόμα και σήμερα δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Παρά το ότι λοιπόν τα τρόφιμα είναι απαραίτητα, παρά το ότι εισάγουμε συνέχεια τρόφιμα, τα εδάφη τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν τα χρησιμοποιούμε για την παραγωγή τροφίμων. Έτσι δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε οι γεωργοί στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Ε, είναι μια απορία την οποία έχουν οι εκλογείς μας. Θα πρέπει οι άμεσες πληρωμές να συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο παράγεται στις εκτάσεις αυτές. Δεν θα πρέπει να πληρώνουμε μόνο και μόνο επειδή ε, φροντίζουμε το χόρτο σε ορισμένες εκτάσεις και δεν παράγουμε τίποτα απαιτείται να είμαστε πιο εφάνταστοι και να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με απλούς τρόπους. Να θέσω και μία επιπλέον ερώτηση σχετικά με την ε, ρύθμιση των πληρωμών. Ίσως, ε, όπως είπα, η κυβέρνηση της χώρας μου να είναι υπεύθυνη γιατί οι άμεσες πληρωμές είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες πληρωμές ε, τις οποίες παίρνουν ε, οι γεωργοί από τις παλαιότερες χώρες. Υποτίθεται ότι ελήφθησαν μέτρα έτσι ώστε αμέσως μετά την ένταξή μας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ακόμα και σήμερα όμως διαπιστώνουμε τις πάρα πολύ σημαντικές αδικίες οι οποίες εξακολουθούν να σοβούν στην γεωργία ανάμεσα στις παλιές και στις νέες χώρες. Εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και έξι σχεδόν χρόνια που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούμε ότι θα υπάρξει μια εξομάλυνση στις πληρωμές προς τους μεν και τους δε. Αλλά παρόλα αυτά ε, και φέτος δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και η αδικία παραμένει. Αν δεν αυξηθεί ο προϋπολογισμός για το κομμάτι της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν αυξηθεί κατά 0,67% είναι σαφές ότι δεν θα επαρκέσουν οι πιστώσεις και είναι σαφές επίσης ότι οι νέες χώρες μέλη που δεν είναι πια τόσο νέες ε, δεν πρόκειται να περιμένουν απονομή δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Νίκολσον έχει το λόγο. Uh, thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε απευθύνω και εγώ, το, το καλώς ορίσατε στην Προεδρεύουσα. Γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι λόγοι της καθυτερημένης αρχής της προσπάθειας, δεν υπήρχε ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα έρθω σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει αναφερθεί ξανά. Στη διάρκεια της Προεδρίας σας είδαμε να ανοίγουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ. Στο πρόβλημα αυτό αναφέρθηκαν και άλλοι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί παράγουν τρόφιμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο διεθνώς. Και αν εξετάσετε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά ε, μέτρα ε, cross compliance τα οποία απαιτούμε να εφαρμόζουν οι γεωργοί μας. Δεν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε τρόφιμα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα τα οποία επιβάλλονται εδώ. Κατά τη γνώμη μου, κανένα τρόφιμο δεν επιτρέπεται να εισάγεται στην Ευρώπη εάν δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρότυπα και προκαλούνται πολύ μεγάλες ανησυχίες από την επανέναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Ένα άλλο θέμα τώρα που έθεσε ο γείτονά μου εδώ σε διάφορες περιπτώσεις για τις διατάξεις που θα εφαρμοστούν από το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ανισότητα ανάμεσα στις χώρες μέλη. Στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία οι γεωργοί που θέλουν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το 40%. Πού βρίσκεται ο ομαλός ανταγωνισμός. Η παραγωγή πουλερικών χρειάζονται όμως τον ομαλό ανταγωνισμό. Και τώρα η επόμενη ερώτηση. Είστε βεβαία ότι το 2012 θα υπάρχει επαρκής παραγωγή αυγών ώστε κάθε ένας καταναλωτής στην Ευρώπη θα θέλει να αγοράσει ένα αυγό να μπορεί και επίσης ότι τα αυγά που θα αγοράζονται δεν θα έχουν παραχθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παλαιές παραδοσιακές συστοιχίες κλοβών ορνήθων και θα, εκεί οι κότες θα έχουν διατραφεί με ε, γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Ο Ζωζέ εγώ βέβαια συμφωνώ πρώτα με τους συναδέλφους μου στα καλωσορίσματα προς την Προεδρεύουσα που ήλθε να κάνει τον απολογισμό. Έχει ξαναέρθει βέβαια σε επιτροπές του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό και έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα λόγω των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά πάντως τούτων λεχθέντων θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου που αμφισβητούν την αξία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρηματά τους, αλλά πάντως η εικόνα που έδωσε αυτή η επανέναρξη δείχνει πόσο η Γεωργία θεωρείται ανταλλακτικό νόμισμα στην πραγματικότητα για να επιτρέπει να πολλούνται ε, υπηρεσίες στις νέες αυτές ε, χώρες. Η Γεωργία εν τέλει αποβαίνει το θύμα, τον, ε, το, το τίμημα πούμε, για να ανοίξουν άλλες αγορές. Το βλέπουμε για τις χώρες Μερκοσούρ, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην παραγωγή βοήου κρέατος στην Ευρώπη και θα είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε την ίδια το ίδιο πρόβλημα όπως με το, με το πρόβιο κρέας πριν από 20 χρόνια και θα σημάνει και το τέλος των πιο ευάλωτων περιφερειών και περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε με τις διαπραγματεύσεις με το Περού, όπου έχουμε κάποιες περίεργες συμφωνίες στη Γεωργία. Παράδειγμα, στην περίπτωση της συμφωνίας με το Περού, προτείνουμε στο Περού να εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζάχαρη, που δεν παράγει όμως, ποιος πταίει, τις πταίει ή ποιος ε, από αυτό. Θα επιμείνω τώρα σε δύο άλλα πράγματα. Μιλήσατε και σωστά είπατε ότι πρέπει να βελτιωθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος της διατροφικής αλυσίδας και το Κοινοβούλιο ψήφισε ε, εν προκειμένου υπό την Προεδρία σας Συνήθω και η ομάδα υψηλού επίπεδου για το γάλα. Το πρόβλημα που βλέπω είναι ότι εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Στην έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου, δεν, ε, από την έκθεση αυτή δεν έγινε τίποτα για να εξασφαλιστεί κάποιο εισόδημα των παραγωγών. Να βγει και να πει ότι οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να απαγορεύσουμε την ε, πώληση με ζημία των γεωργικών προϊόντων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πάμε από κρίση σε κρίση στην Ευρώπη. Και το τελευταίο, αν και δεν έχετε λάβει εσεί ε, την πρωτοβουλία, είναι για το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Είναι τρίτη φορά που μιλάμε γι' αυτό και βεβαίω το θέτω υπόψη σα. Τώρα έρχεται ο κύριο Νταλή, ο Ευρωπαίο Επίτροπο. Ε, σε δική σα Προεδρία, υποθέτω λοιπόν ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας ευθύνεται και αυτό και όχι μόνο της προστασία καταναλωτών. Έχει κάνει μια πρόταση λοιπόν ο Επίτροπος Νταλή να μειώσει το επίπεδο των ελέγχων της ΕΦΣΑ και μας λέει ταυτόχρονα ότι θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να εγκρίνουν αυτές ή όχι την χρήση των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν όλοι οι νομικοί, δεν μπορούν να αντέξουν σε οποιαδήποτε ε, νομική κριτική. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας επιλήφθη, του θέματος αυτού, εάν σε κάποια προσεχή του συνεδρίαση θα επιληφθεί του θέματος αυτού, γνωρίζοντας ότι οι μισές χώρες μέλη της Ένωσης έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα δεχθούν την πρόταση του Επιτρόπου Νταλή. Συγκεκριμένη ερώτηση, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Προεδρεύουσα, σας ε, καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα εδώ. Σας συγχαίρω για, ε, το θετικό απολογισμό της, ε, του έργου στην Προεδρία την τρέχουσα. Στη σημερινή συγκυρία ο Ευρωπαίος αγρότης βάλεται από την οικονομική κρίση, εκτίθεται στην αστάθεια τιμών των αγρατικών προϊόντων, βιώνει αδιαφάνεια και πρακτικές του ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα και καλεί την ανταγωνιστή και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς με αγρότες τρίτων χωρών που παράγουν προϊόντα χωρίς δεσμεύσεις για ασφάλεια και ποιότητα ενώ ο ίδιος δεν έχει κατοχυρώσει την ποιοτική διαφοροποίηση των προϊόντων του έναντι των καταναλωτών. Μάλιστα, με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι έχουμε επιστροφή στο κατακεφαλή αγροτικό εισόδημα στα επίπεδα του 1995. Σε αυτή λοιπόν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που προσπαθούμε χωρίς όμως δυστυχώς ιδιαίτερο αποτέλεσμα να βρούμε τρόπους για την ανακούφιση έστω και προσωρινά των αγροτών επιλέγει η Επιτροπή να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις με την Μερκοσούρ. Η ένταση του προβλήματος φάνηκε και από την πυκνότητα των αναφορών σε αυτό το ζήτημα από πλευράς των συναδέλφων. Ε, είναι βέβαιο ότι μπορεί σε άλλες εμπορικές συναλλαγές να αποβεί αυτή η συζήτηση σε αμοιβαίο όφελος. Είναι όμως βέβαιο ότι στον αγροτικό τομέα ε, τα προβλήματα σε ιδιαίτερους μάλιστα τομείς όπως τα οπορολαχανικά, το βόλιο κρέας, τα πουλερικά ή τα σιτηρά ε, θα πληγούν ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να σχολιάσετε ε, αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και ή δυνατόν να μας ενημερώνατε για τις προθέσεις του Συμβουλίου ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις Επιτροπής για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο Μισελ Νταντέν και μετά η Έγκλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που δώσατε στα θέματα που μας ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξάμηνης προεδρίας σας. Η εισαγωγική σας παρουσία εδώ έφερε πολύ καλά μηνύματα τον Ιανουάριο. Βέβαια, ό,τι συνέβη εν τω μεταξύ δεν σας επέτρεψε να προχωρήσετε απόλυτα καθυστέρησε έτσι και αλλιώς η κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν μέχρι το τέλη Φεβρουαρίου ουσιαστικά η χώρα σας είχε εσωτερικά θέματα αρκετά σημαντικά και αυτό σας απορρόφησε. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουν από την Ισπανική Προεδρία οι γεωργοί της χώρας μου είναι κυρίως η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τους Μερκοσούρ. Το Συμβούλιο ήταν πολύ σιωπηλό μέχρι τώρα στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θυμίζω. Να θυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που δίνουμε δικαιώματα σε εισαγωγικά εισόδου σε παραγωγές από άλλες χώρες, ε, αυτοί οι οποίοι υποφέρουν και οι παραγωγές οι οποίες μειώνονται είναι οι δικές μας. Τι θα κάνουμε με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις σαν παράδειγμα όταν το κρέας το εισάγουμε από τη Λατινική Αμερική οπότε δεν θα έχουμε ζώα να μοβόσκουν εκεί. Λοιπόν, Υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα επίσης ε, με το κλίμα και κάθε φορά που εισάγουμε ένα κιλό κρέας ε, συμπληρωματικά ε, από τη Νότια Αμερική εξαφανίζονται τεράστιες εκτάσεις τροπικού δάσου στον Αμαζόνιο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν ανάμεσα στις ενέργειές μας και ανάμεσα στα λόγια μας. Ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούμε θεσμικά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Υπουργέ να μας μεταφέρετε τελικά και το ποιες είναι οι θέσεις του Συμβουλίου σε ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τον κανονισμό για τα οποροκυπευτικά. Η δική σας χώρα όπως και όλες οι χώρες του Μεσογειακού τόξου θίγονται άμεσα από τον κανονισμό για τα οποροκυπευτικά και το Συμβούλιο σιωπά φυσικά. Η Επιτροπή μας υιοθέτησε εδώ και λίγες μέρες επίσης και μια, ένα έγγραφο προσανατολισμού για την ΚΑΠ. Ε, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει αρκετά μεγάλη συνένεση γύρω από τις προτάσεις αυτές. Θα ήθελα παρακαλώ να μας μεταφέρετε τις αντιδράσεις του Συμβουλίου σχετικά με τους δικούς μας αυτούς γενικούς προσανατολισμούς. Είστε υπεύθυνοι για τη γεωργία και για το περιβάλλον, Υπουργέ. Συνεπώς, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σήμερα για τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων του 2009 για τα εντομοκτώνα. Νομίζω ότι η πρακτική η οποία εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί προβλήματα στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ Μισελ Ελιζαμπέτ Ιέγκλ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και εσάς όλους ιδιαίτερος για τα μικρά πράγματα θα έλεγα τη συνεργασία σας στην προσπάθεια εκπονήσεως της οδηγίας για την προστασία των πειραματόζων όπου μαζί με τις υπηρεσίες σας συνεργαστήκαμε καμιά φορά με κριτικό τρόπο αλλά πάντως συνεργαστήκαμε καλά για ένα δύσκολο θέμα και ευχαριστώ πραγματικά όλους τους συνεργάτες σας στις υπηρεσίες σας. Οι ανησυχίες μας σχετικά με την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική είναι αυτές που σας εξήγησαν οι συνάδελφοί μου προηγουμένως. Εμείς είμαστε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου που επιθυμεί να διασφαλίσει ώστε και το μισό δισεκατομμύριο αυτό Ευρωπαίων πολιτών να έχει στη διάθεσή του επαρκή και καλής ποιότητας τρόφιμα. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι εκεί έχουμε θεσπίσει υψηλά στάνταρτ, υψηλές προδιαγραφές και για την προστασία των ζώων, που δεν τηρούνται παγκοσμίω, ούτε μπορούν και να τηρηθούν, ούτε μπορούν να επιβληθούν παγκοσμίω και αυτό αφορά και τη συνεργασία με τον Μερκοσούρ αλλά και τις διμερείς ε, ε, συμφωνίες με τον Καναδά που μας ανησυχεί όλους τους συναδέλφους μου εδώ και εμένα. Νομίζω ότι πρέπει να πράξουμε πάντα δυνατό και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, ώστε μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Γεωργία να παραμείνει καλή και ανταγωνιστική. Θα σας παρακαλέσω και από εδώ και στο εξή να το λαμβάνετε αυτό ως μέτρο όλων των δραστηριοτήτων σας και για την υποστήριξη των γυναικών της υπαίθρου το θέμα το οποίο έχουμε ε, θεωρήσει εμείς εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικός σε όλους τους τομείς. Έχουμε και έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι όταν θα το συζητήσουμε θα μπορέσετε να τοποθετηθείτε, να θετικά και για τον δεύτερο πυλώνα χρηματοδότησης. Γκλάτενφέλντερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αναλάβατε την Προεδρία σε δύσκολους καιρούς. Δεν μιλώ μόνο για τα αποτελέσματα που μπορούσαμε να επιτύχουμε. Θα θυμούμε την Προεδρία σας για ένα λόγο. Και αυτό θα είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ. Έτσι θα θυμόμαστε την Ισπανική Προεδρία. Πριν από μισό χρόνο, όταν ε, εξηγήσατε το πρόγραμμα της Προεδρίας σας, δεν ενημερώσατε το Κοινοβούλιο ότι προτίθεστε να επαναρχίσετε τις ε, διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ. Εάν το είχατε πράξει, θα είχαμε την ευκαιρία ως Κοινοβούλιο να σας πούμε από την αρχή αυτά που καλούμαστε να σας τα πούμε τώρα, εκ των υστέρων, ασκώντας κριτική στην πράξη σας αυτή. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν αποτυχία, διότι η παλαιά εντολή του 1990 αποτέλεσε την βάση για την επανέναρξη. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει από το 1990 και έχει αλλάξει πολύ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει πολύ. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις αλλαγμένες συνθήκες οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να ξαναρχίσουν στην βάση νέας εντολής η οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη και το γεγονός ότι σε αυτό το μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί, έχει αποκτήσει τώρα 27 πια χώρες μέλη και η νέα εντολή θα έπρεπε να είχε δοθεί όπου να έχει λάβει υπόψη θέματα αλλαγής του κλίματος, παγκόσμια θέματα, συνολικότερα θέματα δηλαδή ε, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των ζώων κλπ η Ισπανική Προεδρία δεν διέθετε ωστόσο αυτή την εντολή και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να διατηρηθούν με την εντολή αυτή. Η κυρία Τότς. Θα ακολουθήσει ο κύριος Γιάρα. Σας ευχαριστώ κυρία Προεδρεύουσα. Τέσσερα-πέντε σχόλια θα κάνω μόνο. Όπως και άλλοι συναδελφοί μου, ανησυχώ ιδιαίτερα από την έλλειψη ελέγχου και κινήσεως της Ισπανικής Προεδρίας στις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Το πρόβλημα που απασχολεί ιδιαίτερα την Βόρεια Ιρλανδία για τους παραγωγούς πατάτας και για την Ιρλανδία και για την ε, Ολλανδία όπου είδαν την παραγωγή τους να μην επιτρέπεται να εισέλθει στο Μαρόκο. Κάτι το οποίο προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στους ε, ε, παραγωγούς αυτούς της περιοχής μου. Και αυτό είναι σημαντικό για τις εσωδίες της επόμενης περίοδου και είναι σημαντικό αυτό για την Βόρεια Ιρλανδία και για όσους αναμένουν εισόδημα από αυτήν τη δραστηριότητα. Επίσης ανησυχώ και εγώ πολύ από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ. Αυτό θα αποβεί καταστροφικό για την ε, Βόρεια Ιρλανδία και ιδίως για την παραγωγή βόλου κρέατος. Πάλι εδώ αφενός σας ακούμε να λέτε ότι συνεργαστήκατε με το Κοινοβούλιο και με την παρούσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά αυτές οι συζητήσεις σας με τις Μερκοσούρ άρχισαν χωρίς πρώτερη διαβούλευση. Και δεν είναι αυτός ο τρόπος συνεργασίας που ε, θεωρούμε εμείς ορθό. Για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και εμείς θέλουμε ισχυρή ΚΑΠ, άρα και ισχυρό προϋπολογισμό, άρα και ισχυρή φωνή απέναντι στο Συμβούλιο. Τέλος, στην Επιτροπή Αλίας όπου συμμετέχω και όπου είναι και άλλα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, ίσως μπορείτε σε κάποια φάση να μας πείτε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και η δική σας σχετικά με την περιφερειοποίηση της ε, πολιτικής αυτής που είναι πολύ σημαντική υπόθεση και που φαίνεται να έχει κάπου αποτελματωθεί μέσα στη γραφειοκρατία που προκάλεσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ κυρία Ντότς. Γεια, ευχαριστώ και για την έλευση σας εδώ και για την διάθεσή σας να συζητήσετε μαζί μας. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια υπόθεση επιτυχίας και όχι μόνο επειδή καταφέραμε να εξασφαλίσουμε παρκή προμήθεια τροφίμων στους Ευρωπαίους πολίτες, είναι επίσης επιτυχία διότι Κατορθώσαμε επίσης οι γεωργοί να δεχθούν να δεχθούν την επιβολή των προδιαγραφών που προκύπτουν από ε, τις επιθυμίες και αξιώσεις των καταναλωτών. Είναι σημαντικό για τους γεωργούς ότι οι προδιαγραφές αυτές οι οποίες ισχύουν και είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της και ο καταναλωτής της θέλει και ο γεωργός της έχει δεχθεί. Θέλει δηλαδή προϊόντα καταναλωτής τρόφιμα τα οποία να έχουν παραχθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο που να είναι ελεύθερα από ορισμένε ουσίες. Συμφωνώ λοιπόν με πολλούς από τους συναδέλφους μου οι οποίοι εξεφράστησαν επικριτικά σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ. Ερωτώ λοιπόν και εγώ πώς σκέπτεστε να λύσετε την αντίφαση αυτή μεταξύ παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισαγωγών. Διότι εν τέλει διακυβεύεται και η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής στα μάτια των Ευρωπαίων παραγωγών. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ, παρακαλώ η Προεδρεύουσα. Εγώ δεν ήθελα να λάβω το λόγο, Πρόεδρε. Γιατί με έχει καλύψει ο κύριος ε, Καπούλος Σάντας, ε, η κυρία Γκαρθία, ο κύριος Μαρτίνεθ. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία ε, με, αγανακτούν και εγώ εργάζομαι στην Επιτροπή Γεωργίας εδώ και 20 χρόνια. Προσπαθώ επίσης να βοηθήσω στην υπόθεση της αναπτυξιακής βοήθειας και ζω στην εποχή μας δεν ζω στο 19ο αιώνα. Φυσικά και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, ότι δηλαδή έχουμε αυτές τις ε, συμφωνίες που αφού γίνουν διαπραγματεύσεις έχουν υπογραφεί. Τέλειωσε, δεν είμαστε ακόμη στις διαπραγματεύσεις. Κλείσανε συμφωνίες. Αυτό που να ότι έχουμε τις υγειονομικές προϋποθέσεις και τις άλλες, οι οποίες ε, είναι αυστηρές όσον αφορά τον έλεγχο των προϊόντων που έρχονται από τον υπόλοιπο κόσμο ως εισαγωγές και ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκρισιμότητα, αντιστοιχεία με τα όσα ισχύουν για τα δικά μας προϊόντα προς τα έξω. Τι γίνεται πρώτα πρώτα, να δούμε τι γίνεται με το Μερκοσούρ. Εδώ άκουσα επανειλημμένα να αναφέρεται ότι δεν υπογράφει συμφωνία με το Μερκοσούρ. Όχι. Απενεπλάκη μια κατάσταση που είχε εμπλακεί πάρα πολύ καιρό. Δεν άκουσα να έχουμε δεξιά ή αριστερή ευρωπαϊκή κυβέρνηση που να μην το χαιρέτησε το γεγονός ότι είχαμε την απεμπλοκή αυτής της καταστάσεως των εμπορικών διαπραγματεύσεων μια σειρά χωρών που όσον αφορά τις ε, συναλλαγές μας αντιπροσωπούν πάρα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα των συνολικών μας συναλλαγών. Επομένω, αυτού του είδου η εμπλοκή ήταν κάτι πάρα πολύ επιβλαβές για την Ευρώπη. Άρα, δεν, είπαμε, δεν λέμε για διαπραγματεύσει, λέμε για απεμπλοκή. Και άρα, τα καταστροφικά σενάρια ανετράπησαν. Και εδώ πέρα έχουμε πέσει μια συνάντηση φάση που με ενισχύουν, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάποιους οι οποίοι πρεσβεύουν την ελεύθερη αγορά, και εδώ και δεκαετίες σηκώνουν λοιπόν αυτό σαν μπαγκέρα ε, και θέλουν πάνω από όλα, την ελεύθερη αγορά. Είναι τα, τα Άγια των Αγίων για αυτούς. Και ξαφνικά, ξαφνικά γυρνάνε και ε, γίνονται προστατευτικοί. Θέλουν τον προστατευτισμό, θέλουν να, να σηκώσουν ένα τείχο, ένα φραγμό, τόσο πολύ. Οπότε Ποιο θα του πιστέψει έτσι. Ούτε οι ίδιοι μπορεί να πιστέψουν τον εαυτό του με αυτά τα οποία λένε και γυρίζουν. Αυτό πάρα πολύ με ανησυχεί. Έχουμε και διάφορου αριστερού συνάδελφου που λένε Να, αλληλεγγύη με τον τρίτο κόσμο. Η σημαία μα αυτό είναι. Για και προσέχτε. Τι θα γίνει. Θα έχουμε εδώ κάποια προϊόντα από χώρε που βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο τραγικό ανάπτυξη και από την άλλη μεριά σύμφωνα με, το, με τη συνθήκη της Λισαβόνας εμείς ήδη έχουμε επιβάλει την βοήθεια την αναπτυξιακή και αυτό να είναι σημαίνει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να υπάρχει μια γενική φλού πολιτική. Αυτό αυτή είναι σημαία μας. Είναι πλατφόρμα μας ιδεολογική. Είναι, το, το, το, το, Ευαγγέλιό μας το να τους βοηθούμε. Επομένως, να, αυτή η συμφωνία με τη Λατινική Αμερική λένε τι κάνει, φέρνει κίνδυνο για κάποια προϊόντα όπου υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία, λέει, να κρατήσουμε στην, στην επιφάνεια κάποιου καλλιεργητέ, κάποιε κάποιες λίγε χιλιάδε ε, καλλιεργητών που ακόμα ασχολούνται με αυτά τα περιθωριακά προϊόντα. Όμως εγώ νομίζω ότι η οπτική μας είναι οπτική μιας αλληλεγγύης και επομένως αυτό και μας, ε, μας προβληματίζει ότι θα γίνει με τη δική μας παραγωγή αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει ε, υψώνοντας κάποιο, κάποιο φρούριο αφήνοντας απ' έξω όλους αυτούς που πεθαίνουν τη πείνας στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι όλα αυτά να τα συγκεράσουμε, να τα συνδυάσουμε και γι' αυτό σας λέω ε, αυτό κάθομαι και υπολογίζω πόσο ε, συνέπεια έχουμε εμεί, σε σχέση με το πόσο συνέπεια έχουν οι άλλοι για την πολιτική που χαράξαμε για την Γεωργία. Αυτά τα οποία έκανε η Ισπανική Προεδρία που μπόρεσε τελικά ε, να καλύψει αυτή μα τη μέρημνα και για τα δικά μα προϊόντα και για τη δική μα Γεωργία αλλά και ταυτόχρονα μπόρεσε να έχει αυτή την ευσυνειδησία, την ευαισθησία τη ελεγγύης που ακριβώ αυτό χαρακτηρίζει εμά του σοσιαλιστές και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους ως Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση είναι πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας και θα δώσω το λόγο εκ νέου στην Ελένα Εσπινόσα για να δώσει κάποιες απαντήσεις σε όλες τις. Την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Σπινόζα. Πρώτα-πρώτα να αρχίσουμε τις απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία τέθησαν. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω εκ προημίου το εξής. Είπατε ότι η Ισπανία είχε εσωτερικά προβλήματα. Όχι. Με τίποτα δεν ισχύει αυτό. Ούτε υπήρχε εσωτερικό πρόβλημα, ούτε υπάρχει. Η Ισπανία έχει ό,τι προβλήματα έχουν και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε δηλαδή αυτήν την διεθνή κρίση. Η διεθνή κρίση έφτασε και στην Ευρώπη, οπότε και εμείς πήγαμε σε θέσπιση κάποιων μέτρων τα οποία δεν διαφέρουν ουσιαστικά ούτε με τα μέτρα που έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Ή τα μέτρα που έχει λάβει η Πορτογαλία, και που ενδεχομένω χρειαστεί να γίνουν και για άλλε χώρες. Επομένω αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και στη συνέχεια να αρχίσω να καλύπτω τι ε, απαντήσεις και τα ερωτήματα που μου θέσατε. Αυτό δε θα πρέπει να το κάνω γιατί όλοι θίξατε πρώτα πρώτα το Mercosur. Τι είπε στην τελευταία παρέμβαση να λάβουμε υπόψη ο κύριος Μαρτίνες. Πρώτη λοιπόν διευκρίνηση ότι δεν ήταν θέμα διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ. Όπως γνωρίζετε με το Μερκοσούρ είχαμε αναστολή, διακοπή των διαπραγματεύσεων το 2004. Το ότι λέμε για διακοπή διαπραγματεύσεων, Για αναστολή διαπραγματεύσεων, αυτό δεν πάει να πει ότι χρειάζεται νέα συμφωνία για να συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις μας. Και βεβαίως χρειάζεται να δώσει το πράσινο φως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για να έχουμε τέτοιες νέες διαπραγματεύσεις. Υποκειμένου δε, τι είχαμε. ακριβώς επειδή έγινε αυτού του είδους η διακοπή, η αναστολή αυτής της διαδικασίας, δεν χρειάστηκε εκ νέου να δοθεί έγκριση από τα θεσμικά όργανα. Οπότε, από το 2004 και μετά δεν είχαμε τίποτα, αλλά ξαφνικά ήρθαν όλα τα προβλήματα πριν από λίγες εβδομάδες. Για να δούμε τώρα. Ποια είναι τώρα η δική μας η, η υποχρέωση είναι το να, να, να, φέρουμε σε αίσιο τέλος αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί πρόκειται για μια αξιόλογη συμφωνία και η συμφωνία είναι αξιόλογη όταν είναι δίκαιη. Δίκαιη σε όλα τα επίπεδα μια που δεν μπορούμε να έχουμε καμία ε, τέτοια ε, στάση που να είναι επιζήμια ή κερδοφόρα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε τώρα να ανοιχτούμε σε αυτή τόσο μεγάλη αγορά με τόσους καταναλωτές πέραν αυτό που είπε ο κύριος ε, Μαρτίνες. Και αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω στα όσα μας είπε. Αυτό σας επισημαίνω. Αυτό έκανα και εγώ ως υπουργό που συμμετέχω στο Σύμβουλο των Υπουργών. Να μην ξεχνούμε ότι αυτό είναι ευθύνη όλων. Είχαμε αυτή τη συμφωνία του 2004. με αρμόδιο το Συμβούλιο το οποίο θα μπορούσε να εγκρίνει μια νέα συμφωνία οπότε και αυτό θα γινόταν με την συναπόφαση. Εγώ δε άκουσα προσχετικά όλα όσα είπατε. Όμως ε, έχουμε κοινή αρμοδιότητα και κοινή ευθύνη. Ό,τι και να εγκρίνει το Συμβούλιο των Υπουργών, διότι αυτό που εγκρίνει το Συμβούλιο εσείς μπορείτε να το, να το καταρρύψετε. Και γι' αυτό σας λέω, μιλούμε για μια τέτοια συμφωνία που θέλουμε να είναι εποφελής για όλους. Δεν θέλουμε κανείς να βγει ζημιωμένος. Πάρα πέρα. Πέρα από το Μερκοσούρ, μου αναφέρατε τα της εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβιότητα και κάποια αντιστοιχεία σε αυτά τα οποία επιβάλλουμε, αυτό που μας επιβάλλουν. Αμοιβιότητα επομένως και επίσης να υπάρχει αυτή η ανιχνευσιμότητα που έχουμε θεσπίσει γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε δίκαιο αποτέλεσμα. Θα συζητήσαμε και ξανασυζητήσαμε αυτά για να δούμε πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί και επίσης είπαμε ότι αυτό θα γίνει μέσω τελειοποίησης των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ό,τι έχουμε, να το αξιοποιήσουμε, να πουλήσουμε τα προϊόντα που έχουμε όσο θέλουμε και να προσέξουμε τώρα ούτω ώστε να πληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που έχουμε τάξει. Τώρα δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία Ακούστηκαν πρώτα το ότι χρειάζεται να υπάρχουν επιστημονικέ μελέτε. Πρόκειται για μια προτεραιότητα. Έτσι θα μάθουμε πώ να ενεργούμε. Και χρειάζεται και να υπάρχει και μια μελέτη για επιπτώσεις οικονομικέ. Και βέβαια η ανάγκη αυτή τη μελέτη δεν έρει το ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν στην συμφωνία με το Μαρόκο. Και η κυρία Γκαρθία μεταξύ άλλων. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε με το πρίσμα της λογικής. Μία προεδρία θα πρέπει να προεδρεύει με πιστικό τρόπο σε ένα συμβούλιο, σε μια ακρόαση, σε μια επιτροπή. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα. Το προβλέπει ο νόμος, κυρία Γαρθία. Ε, είσαστε ευρωβουλευτής. Τι, δε, δεν ήσασταν όμως υπεύθυνοι για αυτή τη συμφωνία, για την κύρωσή της. Μας κατηγορείτε ότι εμείς φρενάραμε τις εξελίξεις για να αποσύσουμε την ευθύνη. Δεν είναι αλήθεια. Προβλέπεται κάποια διαδικασία, προβλέπεται κάποιο timing. Και φυσικά ό,τι να γίνει θα περάσει, θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να, έχουμε, να χτίζουμε παλάτια στην άμμο που να γκρεμίζονται με το παραμικρό. Τώρα, το θέμα αυτό μας παραπέμπει σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία ελέγχθησαν. Πάλι από την κυρία Γκαρθία. Πρόκειται για ισχυρισμού δημαγωγικού σαν για αυτούς που ακούγονται ακριβώς ίδιου ε, στην Ισπανία από το κόμμα της κυρίας ε, Γκαρθία. Ακριβώς τα ίδια χρησιμοποιήσει όπως αυτά που ακούγονται στο ιστορικό της χώρας. έχω να σας πω το εξής. Πολλές φορές γίνεστε αρνητικοί. Αυτά γίνεται με το Λαϊκό Κόμμα που εκπροσωπείτε. Ότι δεν κάνετε να σκεφτείτε ότι η Ισπανία δεν βάζει στο πρόγραμμα το 2020 τη Γεωργία σαν προτεραιότητα. Λέτε δεν, δεν λέει τίποτα αυτό το έγγραφο. Έχουμε αυτέ τι τρει γραμμέ, τρει, πόσε, τέσσερι λέει. Και υποναφέρεται ότι όλε οι κοινέ πολιτικέ και ιδίω η αγροτική πολιτική πρόκειται να συνεισφέρουν στην στρατηγική του 2020 και αναφέρεται ο αγροδιατροφικό τομέα σαν ένα τομέα ανταγωνιστικό, ανταγωνιστικό με κάποιο είδου δυνατότητε, να δώσει μια όθηση στην οικονομία και στην απασχόληση γιατί αυτό είναι η πρώτη μα προτεραιότητα ε, που πρόκειται να είναι η βάση για το, για το, για το, για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρώπης, καθίστε και σκεφτείτε ποια άλλη πολιτική έχει το, το, τόση ποια άλλη παίρνει τόσα, κονδύλια σαν την ΚΑΠ. Μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για στρατηγικό τομέα, μιλάμε για άλλες πολιτικές, παλιές πολιτικές. Για πέστε μας, Πόσες, πόσες αυτές τις πολιτικές ε, έχουν την ίδια κάλυψη, την ίδια πρικοδότηση. Μπορεί να μην σας άρεσε. Εμείς όμως κάναμε το καθήκον μας, κάναμε την υποχρέωσή μας και την κάναμε επί τη βάση μιας συνένεσης. Μας κατηγορείται έστω και συγκαλυμμένα ότι ε, είχαμε συγκεκριμένους ελιγμούς όπως με τη Δανία και, και, και άλλες αναφέρατε. Κοιτάξτε, αύριο η ανταγωνιστικότητα είναι σημείο που θα ζητηθεί στο, στο Συμβούλιο και θα ζητηθεί αυτό η ανταγωνιστικότητα σαν σημείο α, είναι στη μέση διάταξη. Και ποτέ δεν μπαίνει σημείο Α, εάν δεν το έχει προτείνει η Προεδρία και αν δεν υπάρχει συνένεση από όλου. Αυτό σα το λέω, για να ξέρετε όλοι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και προς τα πού κινούμεθα. Κι άλλα αναφέρθηκαν και θα ήθελα να απαντήσω. Εκεί που κάποιος είπε τι έχουν πρώτο ή δεύτερο πυλώνα συγχρηματοδότηση ή όχι. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε την Προεδρία με Επιτροπή ή την Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς έχετε κάποιες αρμοδίες και εγώ έχω άλλες. Εσείς δεν έχει τόσο αρμοδιότητα να διατυπώνετε κάποιες προτάσεις νομοθετικές. Αυτό είναι δουλειά της Κομισιόν. Εσείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να γίνετε, να φροντίζετε για όλη τη, τη, τη σχετική προετοιμασία, ούτω ώστε επί τη βάση αυτής της προετοιμασίας η Κομισιόν να εκπονεί τις πρωτοβουλίες της τις πρωτοβουλίες της, αυτό και το οποίο είχε πει ο Επίτροπος. Ο Επίτροπος που το είπε στα θέματα της ανταγωνιστικότητας και για τα θέματα ισότητας ανδρών γυναικών και όσον αφορά τα γαλακτοκομικά. Οπότε με τέτοιες προτάσεις, ιδέες και πρωτοβουλίες έτσι καταλήγουμε σε κάποιο τελικό κείμενο. ας πούμε η εγγύηση του εισοδήματο. Αυτό το λέει το έγγραφο της Προεδρίας όσον αφορά τη συζήτηση για τη διαχείριση των αγορών. Αυτό υποβλήθηκε και συζητήθηκε στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου και οδήγησε στα σχετικά συμπεράσματα της Προεδρίας. Ούτως ώστε να υπάρχει ένα πιο γενικός προβληματισμό για το μέλλον τη ΚΑΠ μετά το 2020. Και σε αυτή την περίπτωση είπε η Κομισιόν ότι πρόκειται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων όταν έρθει η ώρα για να παρουσιάσει τις πλήρες προτάσεις της. Τις συγκεκριμένες προτάσεις διορθώνει η κυρία Υπουργός. Δεν κατηγορώ κανέναν, το αντίθετο. Η συνεργασία ήταν Πάρα πολύ αρμονική. Και ανέκαθεν οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται με τι δικέ μα υπηρεσίε και έτσι πετύχαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Για πέστε μου. Πότε, πότε πέρασε κάποιο νομοθέτημα σε μηδενική βάση. Μιλάμε τώρα για πενταετία, εξαετία, δηλαδή, λέμε τώρα για το τι θα γίνει το 2013. Μιλάμε για τόσο σύντομη περίοδο. Μιλάμε για τέσσερι μήνε που έχουμε στη διάθεσή μα και που επιπλέον έπρεπε να έχουμε τη συναπόφαση. Πότε έγινε αυτό με οποιοδήποτε κοινοβούλιο. Να, αυτή είναι η πραγματικότητα που είχαμε αντιμετωπίσουμε αυτή στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να ε, δουλέψουμε. Και γι' αυτό και είχαμε την Τρόικα, γι' αυτό και κάναμε τις διαπραγματεύσεις με το κοινό πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια και όχι ρήξη. Η Ισπανική Προεδρία έβαλε τα θεμέλια, η Ισπανική Προεδρία επιτάχυνε τη δουλειά σε όλες τις ομάδες εργασίας, και η Προεδρία κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα. Χαμογελάτε, αλλά κάποια μέρα θα το αναγνωρίσετε. Ότι κατελήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα, τα ομόφωνα. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσει, θα αξιοποιήσει, θα υλοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες. Και άλλα για τώρα αναφέρθηκαν, αυτά τα οποία ε, τέθησαν με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Ο κύριος Νίκολσον, ο κύριος Νίκολσον ε, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα προϊόντα για το τι θα γίνει ε, το 2012. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται αυτά τα προϊόντα να συνεχίσουν να υπάρχουν για τους λόγους που σας προανέφερα. Όμως, άλλος έχει ε, κάτι το οποίο αναφέρατε, αλλά ήδη το έχω συζητήσει με τον Επίτροπο τον κύριο Νταλή. Μου το πεμένα, το είπε και σε συνέντευξη τύπου. Δεν, δεν είναι κουτσομπολιό, δεν λέω ότι κανένα μυστικό. Το είπε συνέντευξη τύπου. Δηλαδή το τι θα γίνει όσον αφορά την, την καλομεταχείριση, την ευημερία, το, το περιβάλλον, σε σχέση με το τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε η κάθε πρωτοβουλία να λαμβάνει υπόψη σε, κάθε κράτος μέλος αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζητήσει. Δηλαδή ότι κάθε φορά που έχουμε κάποια καινούργια μέτρα να υπάρχει κάποια κοινωνικονομική μελέτη η διαφοροποίηση της παραγωγής. Και όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της, ε, του, της ανταγωνιστικότητας. Όταν δουλεύουμε κάθε φορά με βάση κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ο κύριος Μποβέ μίλησε για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σας παραπέμπω σε κάποιες ε, δηλώσεις του κυρίου Μπαρόσο προς το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου 2009. Εκεί δεσμεύθηκε να παρουσιάσει πρωτοβουλία όσον αφορά την νομοθεσία σε σχέση με αυτούς τους, ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ο κύριος Ντάλι ακριβώς αυτό κάνει, ε, υλοποιεί την υπόσχεση Μπαρόσο προς το Κοινοβουλίο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω το τι ε, πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε ως Υπουργείο Γεωργίας για τέτοιου είδους μέλουσα ρύθμιση. Επίσημα ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει αυτή η ευκαιρία μετά από λίγους μήνες. Μετά από τις σχετικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και ε, δική μας ε, συζήτηση με την Βελγική Προεδρία. Προσπάθησα να απαντήσω όσο γίνεται ε, σε όσα μου αναφέρατε τώρα. Προσπαθώ να σας καλύψω σε όλο όσα ζητήσατε, γιατί με τα περισσότερα που είπατε συμφωνώ. Όμως θα πρέπει να δούμε τι έγινε με αυτή την ε, γενική πορεία που αρχίσαμε και δεν πρέπει να την φρενάρουμε. Γιατί η Ισπανία ε, ξεκίνησε σαν πρωτοπόρος ε, σε αυτή την προσπάθεια, όμως τώρα πήραν τη σκητάλη άλλες προεδρίες. Εγώ όλες τις ανησυχίες σας πρόκειται να τις ε, διαβιβάσω αρμοδίως στο Συμβούλιο των Υπουργών, ούτως ώστε να σημειωθεί για όλα όσα αναφέρθηκαν. Όμως πιστεύω ότι μας περιμένουν πολύ σημαντικές προκλήσεις και θα πρέπει μέσω των δημιουργικών προοπτικών να έχουμε μια προετοιμασία επαρκή για την ε, ΚΑΠ. Γιατί έχουμε πει πώς θέλουμε να γίνει η ΚΑΠ. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα τη διαμορφώσουμε και να την κάνουμε ε, ανταγωνιστική και ε, επίσης να, ε, να καλύψουμε και αυτό που ο κύριος Μποβέ για τα γαλακτοκομικά. Όντως, η, τα, τα συμπεράσματα α, καλύπτουν την κατάσταση στα περισσότερα κράτη-μέλη. Όμως θα πρέπει τα συμπεράσματα αυτά του Συμβουλίου να τα κάνουμε κοινοτική οδηγία. Αυτό τώρα απασχολεί τον, τον Επίτροπο Γεωργία, συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επιτρόπους γιατί... De la Άλλωστε δεν είναι καν θέμα Επιτροπής Γεωργίας ε, αυτό το θέμα. Ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε την ε, τελειότητα, αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε όλοι μαζί να το κάνουμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας όσο γίνεται πιο αποδοτική για να πάμε σε αποδοτικότητα, να πάμε σε όσο γίνεται πιο ασφαλή τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Πράγματι σήμερα το απόγευμα μπορέσαμε να ακούσουμε εντελώς διαφορετικές ευαισθησίες και απόψεις και ταυτόχρονα είχαμε μία απάντηση από την κυρία Σπινόζα πολύ συγκεκριμένη τελείωσε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σε πέντε λεπτά ξεκινάει η συνάντηση των συντονιστών.